ισχύει ο διορισμός αυτός θα ισχύσει στα πρακτικά. Η γραπτή δήλωση του 2015 για για την ε, προσφορά ε, ε, τροφίμων που έχουν λήξει και δεν έχουν αναλαθεί προς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις έλαβε 388 υπογραφές. Άρα λοιπόν τις υπογραφές πλειονότητας των μελών του Κοινοβουλίου και βάσει του άρθρου 136 του κανονισμού που συνέταξε αυτή τη δήλωση μαζί με τα ονόματα των, και την δημοσίευση μαζί με τα ονόματα των υπογραφέντων ε, δόθηκαν τα τρόφιμα αυτά στους αποτέλεσμα.